Έχουμε την δήλωση της Αντιπρόεδρου της ε, Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Θα σας παρακαλούσα. έχετε το λόγο. Uh, Πρόεδρε, ε, η κατάσταση ε, στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Ε, η συνεχής αναταραχή και τα σοβαρά κρούσματα βίας στη Βενεζουέλα τις περασμένες εβδομάδες μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Επίσημες πηγές αναφέρονται τουλάχιστον σε 13 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς. Η ύπατη εκπρόσωπος, η αντιπρόεδρος Κάθρι Άστον, ήδη εξέδωσε δύο ανακοινώσεις όπου με σαφήνεια καταδικάζει κάθε πράξη βίας και Ε, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και στην απόφαση του ε, για την χρήση βίας στη Βενεζουέλα. Ο έπατος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε περιστατικά βίας από πλευράς ενόπλων ομάδων κατά αμάχων. Πρέπει να σταματήσει η βία μελητή. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να διατηρήσουν τη δημόσια τάξη και σημειώνουμε την ε, δήλωση του κυρίου Μαντούρο βάσει της οποίας ε, δεν θα ανεχθεί βία η κυβέρνησή του από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ελπίζουμε ε, να μην μείνει στα λόγια αλλά να περάσει και στις πράξεις. Ε, οι διαρκείς ε, δηλώσεις ε, επικριτικές κατά της μίας ή της άλλης πλευράς απλώς οξύνουν το κλίμα που το, ίδιο, το κλίμα αναταραχών που επικρατεί στην κοινωνία και στον πολιτικό διάλογο η κοινότητα των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι ο επίσημος συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Σαντιάκο το 2012 στη Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η Βενεζουέλα μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε σχέση ε, με αδιέρετο των πολιτικών δικαιωμάτων το... η ε, περιπόητες οργανώσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παντός αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις για να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Οι αρμόδιες αρχές ε, καλούνται να διερευνήσουν την υπόθεση σε σχέση με την τύχη των κρατουμένων. Ε, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν νομότυπα κρατούνται, αλλιώς αν δεν αποδειχθεί αυτό θα πρέπει να απελευθερωθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν τάχθη υπέρ ε, της ελευθερίας έκφρασης της απόψεως του συνέρχεστε και τους συνεταιρίζεστε. Οι διαδηλώσεις ε, στην Βενεζουέλα ήσαν πριν από δύο εβδομάδες ε, διότι κατήγηλαν υψηλά ποσοστά εγκληματικότητα, ε, οι φοιτητέ καθώς και σοβαρές ελλείψεις στα πανεπιστήμια. Χιλιάδες άλλοι πολίτες της Βενεζουέλας έκτοτε συμμετείχαν στα συλλαλητήρια λόγω της έλλειψης βασικών αγαθών και του υψηλότατου πληθωρισμού. Ε, βλέπουμε όμως και οπαδούς της κυβέρνησης στους δρόμους ε, του Καράκας. Ε, κανείς δεν πρέπει να κρατείται επειδή ασκεί τα δικαιώματα του, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεστε. Οι δημοσιογράφοι και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να ασκούν αυτές τις ελευθερίες τους ε, ανεμπόδιστα. Ε, υπάρχουν αυθαίρετες πράξεις ε, λογοκρισίας. Το Twitter παραδείγματος χάρη αναφέρει ότι έχει παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε φωτογραφίες. Αλλοδαπή ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί έχουν, έχει απαγορευτεί μάλλον η λειτουργία τους. Δεν, μπορεί να, δεν υπάρχει, δεν κατοχυρώνεται πλέον η ελευθερία έκφραση απόψεων στα ΜΜΕ. Υπάρχουν οικονομικές σοβαρές δυσκολίες. Το ποσοστό του πληθωρισμού έχει φτάσει στο 56%. Η έλλειψη ασφάλειας και εγκληματικότητα ε, γνωρίζει άνευ προηγουμένου επίπεδα ε, ε, το πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πολιτικού διαλόγου θα πρέπει να σε αντικείμενο συμφωνίας με την αντιπολίτευση. Όταν ο πρόεδρος Μαντούρα ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι, στην εναρκτήρια ομιλία του είπε ότι ήθελε να ε, κυβερνήσει ε, όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας ε, ε, χωρίς εξαιρέσεις ε, ήθελε ένα ενωμένο έθνος ε, και ήθελε να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες όμως γνώριζε ότι το 50% σχεδόν των πολιτών είχαν ψηφίσει τον ανθυποψήφιο του και άρα θα έπρεπε να ακούγεται η άποψή τους στο δημόσιο διάλογο. Οι πολίτες της Βενεζουέλας έχουν όλο το δικαίωμα να αποφασίσουν για το πεπρωμένο της χώρας τους. Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να να εισακούσει ε, τις επιθυμίες ε, όλων των πολιτών ε, ναι, για να υπάρξει πολυφωνία στην έκφραση της δημόσιας νόμης. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εμείς, Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάλα Φράγκα. Παρακαλώ. Εχθές συζητήσαμε εδώ στην Ολομέλεια τα φρικτά γεγονότα της Ουκρανίας και στην Ουκρανία υπάρχουν αρκετοί, για την Ουκρανία υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων και εγώ, αλλά και η Βενεζουέλα ε, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες λόγω ε, ετών πολιτικών δυσκολιών. Εσείς αναφέρθηκετε στα, ε, στα περιστατικά βίας, ε, μία... Ε, καταστρεφτική πολιτική για, τα, την οικονομία και υπάρχει ε, και σπάνιδα τροφίμων σε μία από τις ε, χώρες που έχουν τις περισσότερες πρώτες και πετρέλαιο στον κόσμο. Και μάλιστα ε, είναι τόσο δραματική κατάσταση στη χώρα που χρειάστηκε να ε, προσέξουμε τι συμβαίνει ε, στη χώρα αυτή από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε εικόνε παιδιών, νέων ανθρώπων νεκρών στου δρόμου, είδαμε να φυλακίζεται ένα από του ηγέτε τη αντιπολίτευση, είδαμε να υπάρχουν επιθέσει στο Κοινοβούλιο τη Μαρία Κολίνα Ματσάντο, του κ. Ροσάλε, μέλη τη αντιπολίτευση, του οποίου επιτέθηκαν αγρίω εντό του Κοινοβουλίου, με ε, μέλη του τύπου, δημοσιογράφους, ε, τηλεοπτικά κανάλια, το CNN ε, το 24 ώρες, το κολομβιανό κανάλι αναγκάστηκαν να κλείσουν η Βενεζουέλα είναι μια ε, χώρα, κύριε Πρόεδρε, που υποχωρεί, δεν προοδεύει. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μάριο Βαργαζιώσα, ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας και είναι μια χώρα η οποία δεν έχει δημοκρατία, δεν το είπα εγώ, το είπε δύο φορές ο πρόεδρος της Κωνσταντίνα που έχει πάρει Νόμπελ Ειρήνης. Ε, και ε, υπενθυμίσαμε τις προάλλες ε, πόσο μεγάλο θάρρος έχουν επιδείξει οι πολίτες της Ουκρανίας. Όταν επέστρεψα από το Κίεβο ε, διάβαζα το άρθρο ενός εγνωσμένου κύρου που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει θάρρος για να εκφράσουμε την άποψή μας, τις πεπιθήσεις μας, την ελεύθερη γνώμη μας, τη σκέψη μας. Και νομίζω ότι αυτοί οι νέοι, αυτοί οι νέοι οι οποίοι διαδηλώνουν στους δρόμους αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους ε, για να ζητήσουν μια καλύτερη Βενεζουέλα, αυτοί ακριβώς χαρακτηρίζονται από αυτή την άσκηση θάρρους και το κάνουν ε, κύριε Πρόεδρε ως άτομα τα οποία πρεσβεύουν αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και εμείς εδώ στην Ολομέλεια όπως είπε και ο προηγούμενος κάτογος ε, βραβείου Ζαχάρο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουν να τους κυριεύσει ο φόβος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράγκα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκαρσία. Eh, ναι, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, είπαν οι προλαλήσαντες, η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή βυθίζεται στην αβεβαιότητα, στο φόβο, στην αντιπαράθεση και τα τελευταία 15 χρόνια ε, δεν μας αφήνουν να ε, ησυχάσουμε. Ε, επειδή χάθηκαν όλες οι βασικές αρχές, οδηγηθήκαμε σε ειρηνικές διαδηλώσεις και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την βίαιη επίθεση από πλευράς κυβέρνησης και έχουμε ανησυχητικό αριθμό και θανάτων και τραυματιών και ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν φυλακισμένοι. Όλο αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαφορήσει μπροστά σε αυτό το μέγεθος της βιαιότητας ε, απέναντι σε έναν ειρηνικό λαό ο οποίος επιθυμεί το καλύτερο για τη χώρα του και ξέρει ότι μπορεί να το αποκτήσει γιατί είναι μια χώρα πλούσια, έχει κοιτάσματα πετρελαίου και κανονικά θα έπρεπε αυτό να είναι η πηγή της ανάπτυξής του. Αλλά η κυβέρνηση τα χαρίζει σε ε, φιλικές χώρες ε, γιατί θέλουν να είναι θεματοφύλακες ασφάλειάς τους. και υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες μας ζητούν να ε, πούμε δύο λόγια για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλήσουμε γι' αυτό και να υπερασπιστούμε τη μνήμη τους εδώ, διότι ορισμένες φορές ε, θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πόρα απέχει από την έγκριση μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για αυτούς, ε, διότι αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν έχουν στην πραγματικότητα τίποτα άλλο πέραν από εμά. Εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν να τίνουμε χείρα βοηθείας. Υπάρχει παρουσία 30.000 ε, ε, ε, κουβανών πρακτόρων οι οποίοι αποσταθεροποιούν τη χώρα και θα πρέπει να γίνει κάτι. Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι δυνατόν προκειμένου η Βενεζουέλα να γίνει καλύτερη, πιο ειρηνική και πιο σταθερή χώρα. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές παρακαλώ να τηρούν τα χρονικά τους όρια. Η επόμενη ομιλητρία είναι η κυρία Βέμπερ. Για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο λόγος που έχουν ε, ξεκινήσει και έχουν ξεσπάσει αυτοί οι τεράστιε διαδηλώσει στην Βενεζουέλα είναι σαφή. Ε, απόλυτη ελευθερία, ανικανότητα τη κυβέρνηση να προστατεύσει ε, του πολίτε και έλλειψη βασικών τροφίμων. Αντί να φροντίσει το λαό η κυβέρνηση αποφασίζει να αντεπτεθεί. Και αυτό ω τώρα έχει ω αποτέλεσμα 13 νεκρού, πάνω από 70 τραυματισμένου και εκατοντάδε 100 ανθρώπου ε, Και Εκ παραλίλου, ανησυχούμε ιδιαίτερως για την στρατηγική της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση και να, να στείλει την αντιπολίτευση στη φυλακή μαζί με τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσιογράφους, φοιτητές. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της για τα τεράστια σφάλματά της και να δράσει αναλόγως δεν μπορεί να συνεχίσει να κατηγορεί τον κόσμο και να τον θεωρεί ε, ένοχο. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους κόσμους. Καλούμε λοιπόν προς τον ειρηνικό διάλογο να προσπαθήσει να βρει τη μέση λύση, τη μέση οδό προς ε, όφελος του λαού. Εκ παραλλήλου μέλος του Ευρωκοινοβουλίου με ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα του τύπου και της λογοκρισίας της περιορισμένης πρόσβασης στα μπλοκ και τα κοινωνικά μέσα. Πάνω από 60 μέλη του τύπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι θύματα το, της αστυνομίας, της χωροφυλακής και είναι καθήκον της κυβέρνησης να βάλει ένα τέλος σε τέτοιες πρακτικές, να ερευνήσει, να διερευνήσει και να επιβάλλει κυρώσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εξασφάλιση ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και της εύρυθμα λειτουργούσας αντιπολίτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Ταβάρες. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το να ανήκει κανείς σε μια πολιτική οικογένεια δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την, τον απολυταχειρισμό, τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό αυτής της οικογένειας που εκδηλώνεται ορισμένε φορές, διότι εδώ μιλάμε για αστυνομική βία και ορισμένες φορές κατηγορούμε τη δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Στην Κολομβία όταν καταδικάζουμε τις πράξεις βίας δεν μιλάει κανείς από, την, ε, από το Λαϊκό Κόμμα ε, και αντίστοιχα πιέζει η αριστερή πτέρυγα για την έκδοση ενός ψηφίσματος. Ήθελα να σας πω μόνο ότι από την πολιτική μας οικογένεια της αριστεράς υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Αμερικανικός εμπειριαλισμός χρηματοδοτεί ε, τις βιοπραγίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το ίδιο βλέπουμε να λέει η κυβέρνηση της για την αντιπολίτευση, στη Συρία το ίδιο, στην Βιρβανία το ίδιο. Ε, καταλαβαίνετε ότι οι πολιτικές οικογένειες ε, δεν έχουν σημασία. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εδώ στο Κοινοβούλιο είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να θυμόμαστε τι έγινε εδώ στην Ευρώπη, με τη Βουλγαρία, με την Ουγγαρία. Ε, πριν στραφούμε στην Βενεζουέλα και αυτό που πρέπει να ζητούμε είναι να κατοχυρωθεί η ασφαλής διαβίωση όλων των πολιτών της Βενεζουέλας και να διαφυλαχθεί το δικαίωμά του για ειρηνικέ, το τονίζω, ειρηνικέ διαδηλώσει, και το ίδιο επαναλαμβάνω για όλου του πολίτε τη Βενεζόλας. Τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Ε, θα πρέπει να εξαλειφθεί η φτώχεια γιατί αυτή είναι η βασική πηγή των διαδηλώσεων στη Βενεζόλα. Σα ευχαριστούμε, ο κύριο Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι ποτέ δεν ήμουν υπερμάχο του Χιούγκο Τσάβε ε, στην Βενεζουέλα που ήταν ε, όπως ε, και ο Μαντούρο υποστηρίζει τις δικτατορίες. Αλλά αυτό το ψήφισμα δεν έχει να κάνει τίποτα με τις οικονομικές πολιτικές που ήταν καταστροφικές που ακολούθησαν. Ουσιαστικά αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα του κόσμου να διαδηλώνει κατά της κυβέρνησής τους χωρίς αντίπεινα και να εκφράζει την άποψή της με ελεύθερο τύπο και μέσα από το διαδίκτυο. Εγώ από την ομάδα μου ασφαλώς καταδικάζω τους, τις 13 τηλεφωνίες των διαδηλωτών από τις αστυνομίες και αποστέλω συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει έρευνα και να προσαχθούν οι υπέτειοι. Ο Μαντούρα μπορεί να έχει εκλεχθεί δημοκρατικά, αλλά οι πρακτικές τους ενδεχομένω θα βλάψουν ανεπανόρθωτα τα δημοκρατικά διαπιστευτήριά του. Μιλάμε για υψηλά ποσοστά δολοφονιών και τώρα έχουμε ε, ανεξέλεκτες ε, δυνάμεις που στρέφονται κατά των φοιτητών, κατά των διαδηλετών, κατά της αντιπολίτευσης και αυτό ενδεχομένως να σπρώξει τη χώρα στο χείλος του εμφυλίου. Ο πρόεδρος Μαντούρο, ο οποίος ε, έχει αρχισήσει να συμπεριφέρεται όλο και πιο πολύ όπως ο μέντορας του ο Κάστρο στην ε, Κούβα θα πρέπει να απελευθερώσει τους κρατουμένους και να διασφαλίσει ότι οι ομάδες που δρούν ε, από πλευρά της κυβέρνησης θα αφοπλιστούν χωρίς καθυστέρηση και όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει Όλες οι φωνές αυτές θα πρέπει να εισακούονται σε μια δημοκρατική κοινωνία και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να το πράξει για να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ευχαριστώ. Το, την έχουμε δει αυτή την ταινία πολλές φορές. Είναι η ίδια ταινία που είδαμε το 2002 ε, όταν έγινε επίσης ε, το πραξικόπημα που οργάνωσε η δεξιά με τις φασιστικές αμόδους ε, και τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ μαζί με τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν διάφορα ντοκιμεντέρ που το αποδεικνύουν αυτό και δείχνουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από σταθεροποίηση, εγκληματικές ενέργειες που προέρχονται έρχονται από την αντιπολίτευση αλλά και από ομάδε που υποστηρίζουν την κυβέρνηση με τα ίδια όπλα. Ε, θανατώνονται όλοι, καταστρέφονται οι υποδομέ, ε, λείπουν τα βασικά ε, αγαθά. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί πολύ έξυπνο ότι αυτά τα υποκινεί η ίδια η κυβέρνηση τη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει ελευθερία απόψεων, υποκινούνται πράξει βία, παραβιάζεται το Σύνταγμα. Το πρόβλημα είναι ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν καταδικάζει αυτή την οδό που ακολουθεί η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ε, με τα διατάγματα με τα οποία πλέον κυβερνά αντί για το Σύνταγμα. Πρόκειται λοιπόν ε, για μια, ένα πραξικόπημα. Ε, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για αριστερά ούτε για σοσιαλιστές γιατί όλα αυτά υποκινούνται από τη δεξιά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοντή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ζητήσω από τον Επίτροπο να ε, ε, διαβάσει ευχαριστίας μου στην υπατή εκπρόσωπο για τη δήλωση η οποία έγινε. Η Βενεζουέλα είναι μια χώρα ε, με πολιτισμό η οποία δεν αξίζει την κατάσταση αυτή. Ο ένοπλος ε, ε, Ένοπλες δυνάμεις ε, δρούν κατά του λαού. Κύρια ε, συνάδελφοι, υπάρχουν θάνατοι, βασανισμένοι, ε, χωρίς, άνθρωποι που φυλακίζονται χωρίς δίκη. Και ο, η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ελευθερία της. Έχει δίκαιο ο λαός της Βενεζουέλας, αλλά η ελευθερία χωρίς ασφάλεια είναι ανεργία και η ασφάλεια χωρίς ελευθερία είναι δικτατορία. Τον Ιανουάριο του 2013 η κοινότητα των Λατινοαμερικανικών χωρών και της Καραϊβικής αποφάσισαν να υπάρξει ε, μια κοινότητα. Έγινε σημαντικές διαπραγματεύσεις ε, με ε, συμφωνία σύνδεσης με το Μερκοσούρ και ξεκίνησε αυτή η οργάνωση. Αυτή την εβδομάδα υπήρξε σύνοδος κορυφής στη Βραζιλία. Ε, ναι, η Βενεζουέλα είναι μεγάλη χώρα, θέλουμε να έχουμε συνεργασία με αυτή τη χώρα, αλλά πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκόμες στη συνέχεια για ένα λεπτό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 η βία κατά των διαδηλωτών ε, στη Βενεζουέλα οδήγησε σε 50, 50 νεκρούς ε, και ε, χθες το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος Μαντούρο και έχουμε 100 κρατούμενους. Είναι απαράδεκτο. Βλέπουμε τους φοιτητές, τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που καταδικάζουν τον υψηλότατο πληθωρισμό, τα άδεια ράφια, τη διαφθορά, την αυθαιρεσία, την ατιμορρησία, την καταστολή, την κατάργηση των δικαιωμάτων δικαιωμάτων διαδήλωσης, έκφρασης, ε, του συνέρχες του συνεταιρίζεστε, ε, καταδικάζουν ε, την έλλειψη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα τι να σας πω με αυτά που λέτε για την υπεριαλιστική συνωμοσία και το πραξικόπημα. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος όπου όλοι θα συμμετέχουν, ακόμη και αυτοί που είναι δυσαρεστημένοι. Ο αφοπλισμός των ενεπλών δυνάμεων από την κυβέρνηση η καταδίκη της βίας, η διακοπή της δίωξης των δημοσιογράφων, ε, η έγκριση να επαναλειτουργήσουν ε, οι ραδιοτελεοπτικοί σταθμοί που έχουν κλείσει είναι βήματα απαραίτητα για την προστασία του λαού της Βενεζουέλας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπίλαν δεν είναι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Χουντής. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιε είναι οι εξελίξει και η κατάσταση στη βενεζουέλα όχι φυσικά από τα δυτικά μέσα μαζική ενημέρωση διότι παρουσιάζουν τα γεγονότα μεροληπτικά υπέρ τη αντιπολίτευση. ακούστε έφτασαν να ανεβάζουν φωτογραφίε από σκηνέ βία των κατασταλτικών δυνάμεων στην ελλάδα και να ισχυρίζονται ότι αυτά γίνονται στο καράκα. γνωρίζουμε την κατάσταση στην πορτογαλία στη βενεζουέλα από το κοινωνικό έργο που γίνεται δηλαδή μείωση της ανεργίας εξάλληψη του αναλφαβητισμού αύξηση του βιωτικού επίπεδου του λαού γνωρίζουμε από το πολιτικό έργο αγαπητοί συνάδελφοι στη βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. τους δημοκρατικούς κανόνες δεν μπορεί να τους δεχτεί η αντιπολίτευση. στους δρόμους ηγούνται οι χορτασμένοι παιδιά πλουσίων οικογενειών που χάνουν τα προνόμια τους το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο δεν πρέπει να συνενέσει σε αυτή την επίθεση που γίνεται σε ένα κυρίαρχο λαό δεν πρέπει να συνενέσει στην επεκτατική πολιτική των ηπα. είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλα που υπερασπίζονται τις κατακτήσεις και τα κοινωνικά τη δικαιώματα. Ευχαριστούμε Έχετε μία μπλε κάρτα, κύριε Παρακαλώ. Δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βία στο Καράκας και την ε, προκαλεί ο πρόεδρος Μαντούρο. Κύριε Χουντή, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Μα νομίζω ότι έδωσα την απάντηση. Το ότι υπάρχει βία, κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω από ποια χώρα είστε θα ήθελα λίγο να χρησιμοποιήσω και τι δικέ σα εμπειρίε και τι δείχνουν στη χώρα σα τα μέσα μαζική ενημέρωσης. Προφανώ υπάρχει βία υπάρχουν ταραχέ υπάρχουν συγκρούσει, υπάρχουν νεκροί. έχετε ψάξει από πού είναι οι νεκροί; επομένω το ότι υπάρχει βία όλοι το παραδεχόμαστε. το θέμα είναι από πού ξεκινάει προ τα πού αποβλέπει και πώ θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα. και εγώ ισχυρίστηκα ότι η βενεζουέλα είναι μια δημοκρατική χώρα δέχεται μια επίθεση απέναντι στι κατακτήσει το ΔΕΛΑΡ είναι το πετρέλαιο το ομολόγησαν αρκετοί συνάδελφοι το ξέρουμε τόσο καιρό και επομένως το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει να υπερασπιστεί έναν κυρίαρχο λαό που με τη θέλησή του τραβάει έναν δρόμο που ενδεχομένως σε κάποιους δεν αρέσει. Thank you for your answer. Ευχαριστούμε πολύ για την απάντησή σας. Ο κύριος Ματώ Άντρουβερ για ένα λεπτό στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν υποφέρει ο λαός της Βενεζουέλας, υποφέρει και ο λαό των Καναρίων νήσων. Ε, πραγματικά είναι υπονείδευτος ο θάνατος αυτός των ανθρώπων και σήμερα ε, είχαμε και την επέτειο της δολοφονίας του Καρβάγιο που και στη νησιά των Καναρίων πραγματικά ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη φυσικά. Ο λαός της Βενεζουέλας θέλει να ζήσει ειρηνικά και με ελευθερία χωρίς απειλές και χωρίς προβλήματα και αυτό φυσικά έχει δικαίωμα να το κάνει όπως επίσης έχει δικαίωμα να αγοράζει βασικά προϊόντα, να περπατάει στους δρόμους χωρίς να τον δολοφονούν και να μην ε, ε, τον ε, βάζουν φυλακή γιατί διαμαρτύρεται ή γιατί διαδηλώνει ή εκφράζει ελεύθερα την άποψή τους. Υπάρχουν λοιπόν δικαιώματα τα οποία είναι αναγνωρισμένα και δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτά τα επεισόδια με την ατιμορρησία έτσι όπως γίνεται τώρα. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να κοφεύει. Ο λαός της Βενεζουέλας περιμένει τη βοήθειά μας και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Thank you very much ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχω πάρα πολλού ομιλητέ και γι' αυτό λοιπόν θα σα ζητήσω αυστηρά να τηρήσετε το χρονικό όριο του ενό λεπτού. Πρώτο ομιλητές, ο κύριος Κέλαμ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, λύπη μου και την υποστήριξή μου για τι δεκάδε ανθρώπου που έχασαν τη ζωή του. Εκατοντάδε έχουν ε, φυλακιστεί έχουν βασανιστεί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην υπερσκιαστεί η κρίση της Βενεζουέλα από την κρίση στην Ουκρανία. Και οι δύο είναι σημαντικές. Αυτές οι μαζικές διαδηλώσεις αποτέλεσαν μια πιστική αντίδραση στην αυξημένη, στον αυξημένο ε, την έλλειψη βασικών τροφίμων και της καταπάτησης της ελευθερίας της έκφρασης. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση του κ. Μαντούρο θα πρέπει να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τα τραγικά αυτά περιστατικά. Να αφοπλήσει τις ένοπλες ε, κυβερνητικές ομάδες, να απελευθερώσει τους κρατούμενους και να επιτρέψει την ελευθερία εκφράσης και την ελευθερία του τύπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να χαιρετήσω τον ε, πολίτη από τη Βενεζουέλα που είναι εδώ στα θεωρία και να τους καλωσορίσω από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά υποφέρουμε με αυτά που συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα σήμερα ζει μια δραματική κατάσταση και θεωρώ ότι χρειάζεται διεθνή παρέμβαση. Η κυβέρνηση του Μαντόρο ε, δημιουργεί γενοκτονία στη Βενεζουέλα. Πεινάει ο λαό και η κυβέρνηση δεν του επιτρέπει την ελευθερία έκφραση. Δεν ε, επιτρέπει στα μέσα μαζική ενημέρωση και στην αντιπολίτευση να εκφράσουν την άποψή του και του βάζει στη φυλακή. Και αυτή η επαναστατική δημοκρατική κυβέρνηση και βολιβιανή κυβέρνηση όπως αποκαλείται δολοφονεί το λαό της. Ο Μαντούρο και η κυβέρνησή του είναι υπεύθυνοι για αυτές τις βιαιότητες και εμεί, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσουμε την κυβέρνηση Μαντούρο για τα όσα ε, γίνονται και να υποστηρίξουμε το λαό της Βενεζουέλας που ζητά δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία για τη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. η κυρία Μπιλπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι σοβαρή. Έχουμε θανάτους τους οποίους καταδικάζουμε. Ε, εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τα θύματα. Η κυβέρνηση ε, μέσω των κατασταλτικών επιθέσεων και των επιθέσεων κατά της ελευθεροτυπίας ε, είναι επονίδιστη και θα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει πραγματικός αφοπλισμένος και ε, πραγματικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης ώστε να βρεθεί μια ειρηνική, δημοκρατική και συνταγματική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται ο οργανισμός των Αμερικανικών κρατών μπορεί να παρέμβει για να ζητήσει να τηρηθεί ο διαμερικανικός ε, δημοκρατικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αφήσει μόνη της την κοινωνία της Βενεζουέλας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βοηθήσουμε διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινωνικό και οικονομικό χάος και δεν μπορούμε να, σταματή, να σιωπήσουμε, θα πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα στη συζήτηση αυτή να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Ο, Βενεζου... ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Χίγκο Τσάβες, θεωρούσε ότι ο δρόμος για μια καλύτερο κόσμο ήταν ο σοσιαλισμός. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν εκείνοι που όταν πέθανε ο Χιούγκο Τσάβες θέλανε να υποστηρίξουν την εξέλιξη της Βενεζουέλας. Σήμερα στη Βενεζουέλα η κατάσταση, η κοινωνική και η οικονομική διαμορφώνονται πολύ πενιχρή. Η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συναθρίζεστε, η ελευθερία του τύπου, όλες αυτές οι ελευθερίες καταπιέζονται. Θα πρέπει λοιπόν να τα προωθήσουμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Στήρ. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό μια διάβρωση των πολιτικών θεσμών στη Βενεζουέλα και έναν αυξανόμενο απολυταρχισμό λόγω της έλλειψης πολιτικού διαλόγου και των νέων βιοπραγιών κατά των φοιτητών, φαινόμενο απαράδεκτο, η δικαιοσύνη, η πολιτική που ακολουθείται, η κράτηση των ε, φοιτητών ε, είναι αυτά που καταλογίζουν όλοι στον πρόεδρο Μαντούρο. Είχε υποσχεθεί ένα ε, συνέδριο συζήτησης ε, αυτής της κατάστασης, ε, το οποίο τελικά δεν οργάνωσε λόγω έλλειψης πόρων, όπως μας λέει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέριφε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τι θέατρο εδώ στο Κοινοβούλιο. Το δεξιά από τα Ρήγα ανακάλυψε τα δικαιώματα τα ανθρώπινα που τα έχει ξεχάσει στο Ιράκ, στο Μπαχρέιν, στην Κολομβία και τώρα υψώνει το δάχτυλο μαζί με του εταίρους στη Βενεζουέλα, στη ΣΥΠΑ για να πέσει η κυβέρνηση τη Βενεζουέλα. Γιατί, γιατί από τότε που ανέλαβε την ε, πολιτική ηγεσία ο Τσάβες ε, ε, καταπιέζει και απειλεί απειλεί τον φιλελευθερισμό της, ε, των ΙΠΑ και των πολιτικών εδώ σε ό,τι αφορά τα ε, συστήματα που έχουν αυξήσει το βιωτικό επίπεδο των φτωχών στη Βενεζουέλα γιατί έχει εμπνεύσει τον κόσμο σε όλο τον κόσμο έχει εμπνεύσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αλλά δεν θα περάσετε εδώ γιατί το τελευταίο χειρό λοιπόν έχει ε, κατατροποθεί και αυτές οι κινητοποιήσεις από τον κόσμο μπορούν να κινητοποιήσουν μια επαναστατική διαδικασία που θα συμπεριλάβει το τέλος της ιδιωτικής ιδιοκτησίας βασικών τομέων της οικονομίας και του οικονομικού κλάδου μετά από τις εποχές που ζήσαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μέρφυ, από τον κύριο Ταόρες, μπλε Short, please. Yes, Paul. Πολ. Ξέρεις ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο για πολλά ζητήματα, όμως μιλ... είπες ο πασαράν». Ξέρεις πόσο ιερή είναι αυτή η φράση. Είναι οι λέξεις κατά της πολιτικής καταστολής. Πιστεύεις ότι η πολιτική καταστολή που ασκείται από την δεξιά σε εισαγωγικά πλευρά είναι αιτιολογημένη ή πιστεύεις ε, όπως και εγώ ότι η πολιτική καταστολή ε, θα πρέπει να παρεμποδίζεται πάντοτε προς συμφέρον του, της πολυφωνίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών. Απάντησε από τον κύριο Μέρφυ. Δεν ε, πιστεύω πως ε, αυτές ε, οι αντιδραστικές ε, συμπεριφορές τροφοδοτούνται από αυτό το φαινόμενο. Πιστεύω ότι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα προέρχονται από τη δεξιά και ο, ο αμερικανικός υπεριαλισμός έχει παίξει το ρόλο του. Αν δεις ποιοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις είναι οι ελίτ, οι πλούσιοι φοιτητέ. δεν πιστεύω στην καταστολή, πιστεύω στην κινητοποίηση των εργαζομένων για να τροφοδοτήσουν και να προωθήσουν περαιτέρω την επανάσταση. Next is Mr. Kukan for... Ο κύριος Κούκαν ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα καταδεικνύει ότι ένα αυταρχικό καθεστώς δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει. Η βία κατά των πολιτών, η σύλληψη τα εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφθορά, όλα αυτά δεν είναι ενδείξεις μιας χώρας ευημερούσας. Η Βενεζουέλα αλλάζει και αλλάζει από τον κόσμο που δεν βλέπει οποιαδήποτε άλλη διαφυγή από το να ξε, στους δρόμους. Αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων και γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να τηρηθεί η ηρεμία στη χώρα, οι υπεύθυνοι και οι υπέτειοι θα πρέπει να προσαχθούν. Οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα του Μαντούρο θα πρέπει να αντιστραφεί. Θα πρέπει να βρούμε νέους δρόμους, να γίνουν νέες δημοκρατικές εκλογές και να μην γίνουν άλλα επιχειρήματα και πειράματα. Η κυρία, η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά η δημαγωγία και τα ψεύδη που ακούω εδώ πραγματικά με εκπλήσουν. Το 2013 έγιναν εκλογές στη Βενεζουέλα. Δημοτικές, νομοθετικές, προεδρικές, περιφερειακές. Όλες αυτές οι εκλογικές αναμεκρίσεις ε, διοργανώθηκαν δημοκρατικά από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ε, υπάρχει δημοκρατικό αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μία απόπειρα μέσω αποσταθεροποίησης ε, να ε, διαμφισβητήσουμε αυτό το οποίο αποφάσισε η κάλπη. Προσπαθούν να θεωρήσουν ότι το δημοκρατικό κράτος της Βενεζουέλας που έχει κράτος δικαίου και κυβέρνηση δεν είναι σωστό υπάρχει, ε, ε, θέλουν να φτάσουμε στην κατάσταση της Ονδούρας ή της Παραγουέας και αν, γιατί όχι να φτάσουμε και στην κατάσταση της Αιγύπτου σήμερα. Πραγματικά γίνεται μια ε, πραγματική επίθεση κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Ε, κανείς, ούτε ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, ούτε ο Μερκοσούρ, ούτε κανένας άλλος οργανισμός δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ. Ευχαριστώ κύριο Μπιέλεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όλοι το ίδιο θέμα αναρωτιόμαστε και το ίδιο ερώτημα αναρωτιόμαστε. και για το Καράκας και για το Κίβο. Οι διαδηλώσει καταλήγουν σε αιματοχυσία. Και δυστυχώ, οι δυνάμεις της κυβέρνηση χρησιμοποιούν όπλα όπλα κατά των διαδηλωτών. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους ε, διαδηλωτές και θα ήθελα να καλέσω την κυβέρνηση να βάλει ένα τέρμα στη βία κατά των πολιτών και απευθύνω αυτή την έκκληση προς την κυβέρνηση να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα στην ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του τύπου. Η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του Αναμένω λοιπόν πραγματικά επικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Σκέλη. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Βενεζουέλα γιατί έτυχε να έχω ένα αδελφό που είναι εκεί από το 79 Ιεραπόστολε και μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλή αξιοπρεπής οι ε, πολίτες της Βενεζουέλας και αυτό που θέλουν είναι μια ευημερία. Ο Τσάβες τους την έχει αρνηθεί εδώ και χρόνια γιατί είναι πλούσια η χώρα. Δυστυχώς όμως ε, αποκλειστικά και μόνο στην ελίτ πηγαίνουν ε, τα πλούτη της χώρας. Αυτή τη στιγμή ε, ο, ο Μαντούρο δεν έχει το ίδιο χάρισμα με τον Τσαβές και δυσκολεύεται ε, να κυβερνήσει με δημοκρατικά μέσα. Την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της αντιπολίτευσης, την ελευθερία έκφρασης ε, πρέπει να την σεβαστεί και ε, χρειάζεται διεθνής παρατήρηση των επομένων εκλογικών αναμετρήσεων για να υπάρξει τήρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και προστασία της ελευθερίας όλων και κυρίως ανύψωση των συνθήκων διαβίωσης των μη εχόντων Κυρίω επειδή πρόκειται για μια ε, χώρα με πλούσιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Ε, ευχαριστώ, ε, συγγνώμη κύριε Μέρφυ, αλλά δεν έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε και για τι καταληκτικέ παρατηρήσει, θα δώσω πάλι το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα εν είδη συμπεράσματος να επαναλάβω τα βασικά σημεία της προηγούμενης παρέμβασής μου. Ε, η χρήση βίας ε, και η μυσαλλοδοξία είναι τα βασικά φαινόμενα στη Βενεζουέλα, οι διαρκείς αναταραχές, οι τραυματισμοί ε, και οι κρατήσεις φοιτητών και ε, πολιτικών ακτιβιστών είναι πάρα πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι εθνικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε να ασκείται ελεύθερα η ελευθερία του συνέρχεστε και η ελευθερία της έκφρασης όλων των πολιτών της Βενεζουέλα η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος των δημοσιογράφων. Ε, όλοι οι πολίτες ε, θα πρέπει να μπορούν να εκφράζονται ε, σε πολυφωνικά ΜΜΕ. Είναι νόμιμη, νόμιμο το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά. Ε, και θα πρέπει να ενταθεί ε, ένας διάλογος όπου θα ακούγονται όλες οι φωνές με τρόπο ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα βίας. Ευχαριστούμε. Έχω λάβει έξι σχέδια ψηφίσματος για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Η κοινή συζήτηση λίγη τώρα και η ψηφοφορία των ψηφισμάτων θα γίνει σήμερα στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε διάφορα κράτη-μέλη.